Η μερίσια διάταξη ε, μας επιβάλλει την εξέταση της έκθεσης Κοφεράτη σχετικά με την πρόταση οδηγίας ε, για την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και μια στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχήν τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης. είναι πραγματικά αυτές οι ευχαριστίες μου είναι πραγματικές και όχι τυπικές, γιατί η διαδικασία ήταν πολύ μακρά. Ε, καταρχάς, ε, αναβάλαμε την ψηφοφορία στην Επιτροπή. Εν συνεχεία ψηφίσαμε και στείλαμε το κείμενο στην Ολομέλεια μαζί με μια απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων. Η ψηφοφορία προβλεπόταν για τον Ιούνιο στην, ε, στην Ολομέλεια και τελικά είπαμε θα ψηφίσουμε τον Ιούλιο και αύριο τελικά ψηφίζουμε. Καθυστερήσαμε. Αλλά νομίζω ότι μια λογική επιλογή μας επέτρεψε να εμβαθύνουμε την ουσία της στην ουσία της πρόταση για περίπλοκα αμφιλεγόμενα θέματα όπου πολύ λογικό είναι να έχουμε απόψεις αποκλίνουσες. Χάρη στους σκιώδεις εισηγητέ, χάρη στον εισηγητή της ΕΚΟΝ που τον ευχαριστώ, ε, φτάσαμε εδώ. Πριν μπω ε, εντάχει στο περιεχόμενο της οδηγίας, θέλω να πω κάτι στην Επιτροπή. Εγώ θεωρώ αυτή την οδηγία ως ένα πλαίσιο πολύ πιο ευρύ. Πρέπει να καθορίσουμε ε, με πιο γενικό τρόπο το προφίλ της διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών εταιριών. Ε, ξεκίνησε ο Ζακ Ντελόρ με ένα κείμενο το 1993. Εμείς ε, συνεχίζουμε στην κατεύθυνση που μας υπέδειξε. Είναι μια δύσκολη δουλειά, αρκετά θετική όμως και σήμερα ασχολούμαστε με τους shareholders, με τους ε, μετόχους. Εν συνεχεία θα περάσουμε στους stakeholders για να δώσουμε μια κοινωνική διάσταση στην ε, επιχείρηση που θεωρεί ότι είναι στοιχείο αναφοράς η Πρόεδρός μας. Γι' αυτό λοιπόν περιμένω περαιτέρω πρωτοβουλίες από την Κομισιόν προς αυτή την κατεύθυνση που σας ανέφερα. Τώρα, όπως σας είπα, φτάσαμε στο να καθορίσουμε το μακροπρόθεσμο προσανατολισμό των επιχειρήσεων και των μετόχων και να αυξήσουμε τη διαφάνεια για βασικά στοιχεία της διαχείρισης των επιχειρήσεων ή της διακυβέρνησης, της λεγόμενης εταιρική διακυβέρνησης. Συμφωνήσαμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να ταυτοποιούν του ε, μετόχου του και μιλάω για τι συγμένε στο χρηματιστήριο ε, επιχειρήσει. Προβλέπονται μέτρα για τη βελτίωση τη δυνατότητα άσκηση του δικαιώματο ε, ψήφου από του μετόχου, που είναι στοιχείο και δημοκρατικότητα αλλά και αποτελεσματική διαχείριση οποιασδήποτε επιχείρηση. Επίση, η διαβίβαση των πληροφοριών σε όλου του ενδιαμέσου θα καταστήσει πολύ πιο αποτελεσματική την δουλειά των μετόχων, αλλά και θα γίνεται με τα γνώσεως η δουλειά αυτή. Επίσης, ε, κάποια μέτρα, αν εφαρμοστούν σωστά, θα αυξήσουν τη διαφάνεια μεταξύ των θεσμικών επενδυτών, των ε, διευθυντικών στελεχών και των ε, συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Γιατί αν υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή, οι επιχειρήσεις θα ξέρουν πολύ καλά τι έχουν να περιμένουν ε, οικονομικός πώς, ε, μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Υπάρχουν επίσης ε, άλλα μέτρα για την αύξηση της διαφάνειας των λεγόμενων advisor, των συμβούλων. Επίσης εδώ είπαμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις διαφάνειας τις επιβεβαιώσαμε και εμείς αυτές τις επιλογές της Κομισιόν για τα στοιχεία της διαφάνειας. Το ίδιο ε, σημαίνει και για τις ε, συναλλαγές που θα πρέπει να υφίστανται σε υπόκειται σε ελέγχους και θα διαφοροποιούνται ανάλογα με την νομοθεσία που ισχύει σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωση όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείε. Ε, οι αλλαγέ που προτείνουμε εμεί θα μα επιτρέψουν να λάβουμε υπόψη αυτέ τι εθνικέ ιδιαιτερότητε, χωρί οι ιδιαιτερότητε αυτέ να θέσουν αμφιβόλο την τον ενιαίο χαρακτήρα των ευρωπαϊκών πολιτιών. Επίσης, οι, οι διαχειριστές συγγνώμη, περιουσιακών στοιχείων. Ε, το είχαμε συζητήσει, είχαμε διαφορές, ε, τελικά βρήκαμε την λύση. Οι μέτοχοι θα ψηφίσουν, αλλά η, ψήφη του, η ψήφος τους θα είναι δεσμευτική ή προαιρετική, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα παίρνει κάθε χώρα. Δηλαδή μπορεί να έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, όχι υποχρεωτικό. Και επίσης ε, η καταπολέμηση της ε, φοροδιαφυγής. Ε, αυτή πρέπει να γίνει μέσω της χρήσης νέων εργαλείων. Ετήσια λογοδοσία για τις εισηγμένες το χρηματιστήριο εταιρείε. Είχα μια εταιρεία, μια έκθεση που είχε μιλήσει στο παρελθόν γι' αυτό. υπάρχει και η οδηγία για τους μετόχους και είναι βασικό στοιχείο νομοθετικού χαρακτήρα ε, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά, τα προβλήματα που είχαμε. Ευχαριστώ όλους όσους ε, άκουσαν και θα ακούσω με μεγάλο ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ. Η Γιούροβα, η κυρία Γιούροβα, η Επίτροπος από την Επιτροπή. Ευχαριστώ, αξιότιμοι βουλευτέ. Ε, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείχνετε για αυτή την πρόταση. Θα ήθελα να σα επιθυμίσω εν συντομία ποια ήταν η πρόθεσή μας όταν υποβάλαμε αυτή την πρόταση. Θυμήστε ότι έπληξε η χρηματοοικονομική κρίση, την παγκόσμια οικονομία και τις κοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα σφοδρά. Η Βλέπουμε τις δομές ε, της οικονομικής διακυβέρνησης πιο ξεκάθαρα και έχουμε την εντύπωση ότι ε, ε, ήταν βαθύτερη και τρονότερη η κρίση λόγω των παραμέτρων που ρυθμίζονται μέσα σε αυτή την πρόταση. Προσπαθήσαμε λοιπόν μέσα από αυτή την πρόταση να καλύψουμε τις ατέλειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτω ώστε να επιστρέψουμε στην μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια οι κεφαλαϊκές αγορές καθοδηγούνταν από επενδυτικά παιχνίδια και όχι από καλά σωστά ενημερωμένη επενδυτική πολιτική. Ε, το ίδιο συμβαίνει και στα στεξιδωτικά κεφάλαια. Ο στόχος τους είναι να έχουν μακροπρόθεσμες καλές ε, ε, επιδόσεις, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν πιέσει τις εταιρείες βραχυπρόθεσμα επενδύοντας ακριβώς σε αυτές τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Εμεί χρειαζόμαστε όμω πιο μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και πιο μακροπρόθεσμη συμμετοχή των μετόχων. Χρειαζόμαστε λοιπόν ανταγωνιστικότερε επιχειρήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύουμε ότι ενισχύοντα την οικονομική εταιρική διακυβέρνηση θα έχουν οι επενδυτέ, τα απαιτούμενα μέσα ούτω ώστε να μπορέσουν να προσπα... προστατεύσουν ε, τα συμφέροντά του και καθιστώντα έτσι και ελκυστικότερε ευρωπαϊκέ επιχειρήσει για του επενδυτέ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κομφεράτη αλλά και όλους για τι προσπάθειε που έκαναν ώστε να προσδιορίσουν επακριβέστερα τη θέση του Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με το συνομοθέτη. Θα ήθελα τώρα να εκφράσω διάφορες απόψεις σε σχέση με τις τροπολογίες που έχετε καταθέσει. Για τις υποχρεώσεις διαφάνειας, ε, για τα tax rulings, ε, τις φορολογικές ε, αποφάσεις και την, την υποβολή εκθέσεων αναχώρα. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να καταπολεμήσει τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, επιδιώκοντας αποκάλυψη περισσότερων πληροφοριών σε σχέση με τις εταιρικέ επιδόσεις. Τον Ιούνιο ξεκίνησε διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εναλλακτικέ λύσεις, οι οποίες σε θα τροφοδοτηθούν μέσα στην αξιολόγηση αντικτύπου και θα μας οδηγήσουν στο πέρας της διαδικασίας το 2016. Δεύτερον, τα μέτρα σε σχέση με τα κίνητρα για την αυξημένη μακροπρόθεσμη συμμετοχή των μετόχων για τα δικαιώματα ψηφοφορίας αλλά και για τα μερίσματα. Παρότι συμφωνούμε με τους γενικότερους στόχους, το θέμα είναι με ποιο τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε την υλοποίηση αυτών των στόχων, μη αποθαρρύνοντας τους επενδυτές, ε, κυρίω όταν μιλάμε για τις ξένες επενδύσεις, ε, για τους αλλοδαπού επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε ευρωπαϊκές εταιρείε. Δεν πρέπει επίση ε, να ξεχνούμε ότι υπάρχουν και μειοψηφικοί μέτοχοι και έχουν διαφορετικά συμφέροντα. Στη συνέχεια, σε σχέση με τι ε, συναλλαγέ ε, των συμβαλόμενων μερών, γνωρίζετε ότι οι προτάσει που υπήρχαν στο αρχικό μα κείμενο εξασφαλίζουν ένα εναρμονισμένο κατόφλι για την εφαρμογή των αποφάσεων για τι συναλλαγέ των σχετικών μερών. Βλέπουμε ότι το 40% των μετόχων λειτουργούν σε διασυνοριακή βάση και άρα χρειαζόμαστε ενιαίο ορισμό για τα συνδεδεμένα μέρη, αλλιώς ε, δεν θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τον κατακαιρματισμό και το αυξημένο κόστος τόσο για τους ε, επενδυτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστούμε κυρία Γιούρεβα, τώρα ο κύριος Λούντβικσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικά τα μέτρα που τώρα εξετάζουμε ε, και σωστά τα λέτε ότι χρειαζόμαστε τόνωση των επενδύσεων ούτως ώστε να μπορέσουν όλοι βράχοι μακροπρόθεσμα να ενισχύσουν τη δραστηριότητα αυτών των επιχειρήσεων στις οποίες επενδύουν. Όμως ταυτόχρονα σημαντικό είναι ε, να ενισχύσουμε την ενεργό συμμετοχή των μετόχων σε διασυνοριακή βάση. Αυτή την δέσμευση προσπαθεί να προωθήσει το πακέτο το της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως και για τις μικρές επιχειρήσεις πέρα από τις μεγάλες. Υπάρχει υποστήριξη στο Κοινοβούλιο για να αυξήσουμε την διαφάνεια, κυρίως για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν διασυνοριακά. Το να διευρύνουμε τώρα τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων αναχώρα σε άλλους τομείς χρειάζεται μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε να έχουν καλύτερη ενημέρωση οι μέτοχοι για τα όσα συμβαίνουν στην επιχείρηση και επίσης καταπολέμηση της διαφθοράς, της φοροαποφυγής, φοροδιαφυγή και επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Αυτό το θέμα το προωθεί ούτω ή άλλω στους επικείμενους τριλόγου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λούτριξον. Τώρα από πλευρά τη Επιτρο... της Οικονομικής Επιτροπής. Οι εκπρόσωποι των ε, πολιτικών ομάδων. Ζιεύκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Συχνά μιλάμε για τα θέματα αυτά, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Και είναι ενδιαφέρον συζήτηση όχι μόνο λόγω του περιεχομένου της έκθεσης, αλλά υπάρχουν μια σειρά από ερωτήματα κλειδιά που μπορούμε να θέσουμε ιδιαίτερα λόγω των νέων νομοθετημάτων για την εταιρική διακυβέρνηση και άλλα συναφή που θα επιχειρήσουν να ρυθμίσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων εντός της ενιαίας αγοράς. Οπότε το ερώτημα τίθεται εάν ε, θα δημιουργήσουμε καλού επίπεδου θέσεις εργασίας για τους πολίτες μέσω αυτών και πώς θα αντιμετωπίσουμε τους επενδυτές και τους επιχειρηματίες. Θα τους θεωρούμε ε, εκμεταλλευτές και ανθρώπους που θέλουν να ε, κάνουν απάτες ή θα τους θεωρήσουμε διαφορετικά. Ή θα επιχειρήσουμε δηλαδή να είμαστε επικοδομητικοί και να κάνουμε τέτοιες ρυθμίσεις που να μην παρεμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη, αλλά αντίθετα θα τις δώσουν κίνητρα. Θα δημιουργήσουν αυτή την ε, τόσο ε, θρυλούμενη οικονομική ανάπτυξη. Η ελεύθερη αγορά πρέπει επίσης να είναι ένα άλλο ε, στοιχείο κλειδί Ποιο θα δημιουργήσει νέε θέσει εργασία, η Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι. Ε, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, ε, οι ενεργοί επιχειρηματίες ε, δημιουργούν θέσει εργασίας και όπως ξέρετε 95% των επιχειρήσεων μας είναι μικρομεσαίες. Δεν μπορεί να τις αντιμετωπίζουμε καχύποπτα. Δεν μπορεί να θεωρούμε ότι είναι απλώ εκμεταλλευτέ. Και πρέπει να δούμε και το θέμα της αμοιβή ε, των ηγετικών στελεχών. Οι μέτοχοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν πώς θα αμοιχθούν οι μάνατζερ και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, των εταιριών, με βάση και τους στόχους ε, που θα έχουν καθοριστεί και πόσο θα έχουν επιδευχθεί. Χαίρομαι με αυτή την έκθεση και ευχαριστώ και τους συναδέλφους από την Επιτροπή μας, διότι μετά από αναλυτικές συζητήσεις αποφασίσαμε αυτό το κείμενο και αυτό το κείμενο σήμερα μπορούμε να το αξιοποιήσουμε στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Φυσικά δεν θα είναι εύκολες αυτές οι διαπραγματεύσεις, υπάρχουν ακόμη διαφορές, αλλά είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι αν καθορίσουμε σαφώς τους στόχους μας, εάν ε, αναλάβουμε πρωτοβουλίες, θα τα επιτύχουμε, όπως όλοι επιθυμούμε. Ο κύριος Ρέγνερ. Η κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Κοφεράτη. Θαυμάσια εργασία έχει επιτελέσει σε μια κατάσταση που σίγουρα είναι πολύ περίπλοκη. Και το σχέδιο οδηγίας διαμορφώθηκε και βελτιώθηκε μετά από επικοδομητική συζήτηση και με τους ε, σκιώδεις. Εμείς ως Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων νομίζω ότι επιφέραμε αλλαγές, ούτως ώστε να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια για την εταιρική διακυβέρνηση και για την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας. Και θέλω να τονίσω, να τονίσω το ρόλο των σοσιαλδημοκρατών, διότι καταφέραμε σημαντικές πληροφορίες για τη φορολογική στρατηγική και για τον κίνδυνο ορισμένων επιχειρηματικών πρακτικών και για την αμοιβή των ε, ηγετικών στελεχών, όπως είπα, να υπάρχει διαφάνεια σε όλα αυτά. Όμως, ε, κυρία Επίτροπε, υπάρχουν κάποιοι βουλευτές του ΕΛΚ και των φλερευθέρων, που πρέπει επίσης να προσέξουν. Χρειαζόμαστε περισσότερη συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Από ό,τι ξέρουμε, η Γενική Συνέλευση πρέπει να αποφασίζει τουλάχιστον μια φορά κάθε τρία χρόνια να αποφασίζει για τις ε, αμοιβέ των ηγετικών στελεχών. Αυτό ενισχύει τις ε, δυνατότητες συμμετοχής των μετόχων, αλλά αυτό σημαίνει ότι άλλοι εμπλεκόμενοι και εργαζόμενοι δεν συμμετέχουν επαρκώς. Αυτοί όμως ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την επιτυχία της επιχείρησης. Γι' αυτό η ομάδα μας έχει υποβάλει τροπολογίες για να ενισχυθεί ο ρόλος των απασχολουμένων ε, στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Το κείμενο λοιπόν, όπως εγκρίθηκε, περιέχει κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ιδιαίτερα λόγω και των εργασιών μα στην Επιτροπή Τάξε τα μέτρα που θα καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή. Όπως ανέφερε και η κυρία Επίτροπος και πολλοί άλλοι, και ίσως τον και άλλοι, οι εκθέσεις αναχώρα είναι τόσο σημαντικές, ούτω ώστε να μπει φως επιτέλους, να, να ρίξουμε φως στο σκοτάδι. Πρέπει λοιπόν ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αυτή η ρήτρα διότι η αναχώρα δημοσιοποίηση των αναγκαίων πληροφοριών είναι απόλυτα ουσιώδες αίτημα της ε, ομάδας μας. Είναι θέμα της υπόλοιψης της επιχείρησης. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό διακυβεύεται. Διακυβεύεται, συγγνώμη. Και πιστεύω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα όσο δυνατόν περισσότερο. Σήμερα νομίζω ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για να καταπολεμήσουμε τους φορολογικούς παραδείσους και πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Προσπαθώ να είμαι διαλλακτικός, αλλά παρακαλώ να μην καταχράσετε της ε, διαλλακτικότητας αυτής. Παρακαλώ να μην ξεπερνάτε το χρόνο χρονομιλίο σας, ο κύριος Μέσσερ Σμιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σίγουρα χρειαζόμαστε ίδιου κανόνε για όλε τι επιχειρήσει, όμω η πρόταση που έχουμε επιτάπητο ε, υπερβαίνει αυτά τα όρια. Ε, οι προτάσει που κάνουμε υπερβαίνουν τα όσα εμείς ως κοινοβούλιο οφείλουμε να επιδιώκουμε για τι αμοιβέ των διευθυντικών στελεχών, λόγω χάρη ή άλλα απίστευτα ω προ την των επιχειρήσεων. Κατά την άποψή μου, η πρόταση αυτή βασίζεται σε μια συλλογιστική όπου οι εισηγμένε στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις πρέπει να έχουν βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους ως προς τα αποτελέσματα που πετυχαίνουν. Στην Δανία έχουμε επιχειρήσεις που δείχνουν ότι μπορούμε να τις εμπιστευόμαστε μακροπρόθεσμα. Σήμερα όμως την έκθεση ως έχει δεν μπορούμε να τη στηρίξουμε. Θα απόσχουμε. Διότι πρέπει να έχουμε ένα σωστό πλαίσιο, αλλά εδώ υπερβαίνουμε τα απαραίτητα όρια. Ευχαριστούμε η κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοφεράτη και όλους τους άλλους συναδέλφους για τη σκληρή τους δουλειά και την αγαστή συνεργασία που είχαμε για να βελτιώσουμε αυτή τη σημαντική νομοθετική πρόταση. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που μπορέσαμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις στο επίκεντρο, στην καρδιά μάλλον αυτού του κοινοβουλίου, που, προτάσεις που μπορεί να φέρουν κοντά και σε σύγκληση τις προοδευτικές και υπέρ της Ευρώπη ε, δυνάμει. Έπρεπε βεβαίως όλοι να κάνουμε παραχωρήσεις και αυτό έγινε σε πνεύμα συμβιβαστικό σε πολλά σημεία τα οποία πιστεύω ότι δίνουν ένα τελικό αποτέλεσμα που μπορεί να είναι αποδεκτό από όλους μας. Για την ομάδα των φιλελευθέρων είναι καθοριστικής σημασίας η οδηγία αυτή να βελτιώσει την ικανότητα των μετόχων να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στις διασυνοριακές ε, συναλλαγές και να μην προστίθεται γραφειοκρατικό άχθος εκεί που δεν χρειάζεται. Διότι ας το αποδεχτούμε. Οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες και οι εταιρείε δεν θα ακμάσουν επειδή θα προβλέψουμε επιπλέον κανόνες προς μόρφωση Αλλά εάν δημιουργήσουμε ένα καλό επιχειρηματικό περιβάλλον όπου μπορούν να επικεντρεθούν στις βασικές τους ε, ε, αρμοδιότητες. Δεν μπορούμε να παράγουμε μακροπρόθεσμη διάθεση στους επιχειρηματίες να επενδύσουν με ε, επαχθείς νομοθετικές προτάσεις ή χωρίς να δίνουμε φορολογικά κίνητρα. Οι μέτοχοι χρειάζονται πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες αλλά θα πρέπει να αναλάβουν και την ευθύνη να μπορούν να χειριστούν την εταιρεία την οποία διευθύνουν. Εφόσον αυτό δεν προβλέπεται επισήμως, εφόσον αυτό δεν το σχεδιάσουν οι πολιτικοί, ε, θα πέσουμε στα χέρια των γραφειοκρατών. Νομίζω λοιπόν έμφαση σωστά δίνεται από τις προτάσεις της Επιτροπής να ζητάτε μια λεπτομερής πολιτική για την μισθοδοσία και επίσης ε, υποβολή εκθέσεων για τις αμοιβέ των διευθυντικών στελεχών. Δύσκολο να μην καταλάβουμε ή λαϊκιστικό βεβαίως κάπως το μέτρο και θα μπορούσα να δεχτώ ακόμα και περισσότερα, αλλά τελικά η συμβαστική πρόταση σεβάστηκαν τα βασικά σημεία στα οποία υπήρχαν διαφωνίε και προβλήματα. Σήμερα αισθάνομαι πολύ περισσότερο ικανοποιημένη και ζητώ από την ομάδα μου να στηρίξει την συμβαστική πρόταση ε, για να έχουμε την τελική μορφή τη έκθεση και να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε στου τριμερεί διαλόγου και να ολοκληρωθεί αυτό ο φάκελο. Θέλουμε μια οδηγία που να επικεντρωθεί στου σωστού στόχου και στα συμφέροντα των μετόχων παρά στι υποχρεώσει του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαστάλικα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε. Έχουμε σήμερα να κάνουμε με την αναδιατύπωση δύο οδηγιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου. Ένας από τους στόχους είναι να ενθαρρύνουμε τη μακροπρόθεσμη ενεργό συμμετοχή των μετόχων και των επενδυτών. Οι τα διοικητικά στελέχη πολλές φορές ενθαρρύνονται από τους μετόχους να αναλάβουν υπερβολικά ρίσκα για την επίτευξη όμως βραχυπρόθεσμων κερδών. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερο άνοιγμα στις επιχειρήσεις με τη δημοσίευση των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων στις ε, ιστοσελίδες ε, των εταιριών. Αναφέρεται επίσης για πρώτη φορά σε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ζήτημα των αποδοχών ε, των διοικητικών στελεχών. Μας ενδιαφέρει πολύ και το θέμα των εκθέσεων αναχώρα είναι μια σημαντική, ένα σημαντικό μέτρο για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ευχαριστώ πολύ Κύριε Πρόεδρε, με αυτή την πρόταση τροποποίησης της οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι ε, μακροπρόθεσμες επενδύσεις ε, να τις συμπεριλάβει σε αυτό το πεδίο και αυτό είναι εξαιρετικό γιατί η ευρωπαϊκή οικονομία υποφέρει από ε, των επιγουσών καταστάσεων. Το να λάβουμε υπόψη όπως κάνετε και όπως έχετε προτείνει όλους τους ενδιαφερομένους και τους μικρομετόχους αλλά και τους μισθωτούς που είναι και ο πλούτος των επιχειρήσεων. Εξαιρετική πρόταση δεν αρκεί όμως. Ε, χρειαζόταν να προχωρήσουμε περαιτέρω για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτής της αδιαφάνειας ε, που καλύπτει με ένα πέπλο ε, τις δραστηριότητες και συναλλαγές των μεγάλων τέρων και μεγάλων ομίλων. Οι οικολόγοι τόνισαν ε, το ζήτημα της ανάγκης διαφάνειας και έχουμε και τα μέτρα του φορολογικού, επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού που ήθελαν επίσης εκεί να έχουμε πρόοδο. Το σκάνδαλο Lux Leaks νομίζω κατέδειξε σε όλες και όλους ότι ο κόδωνας συναγερμού που είχαν κρούσει οι ιδίως οι οικολόγοι εδώ και χρόνια, πραγματικά ε, μας υποχρέουν να δώσουμε απαντήσεις. Και γιατί, διότι αυτή η περιβό, αυτός ο περιβόητος ε, επιθετικός φορολογικός ε, σχεδιασμός πλήττει άμεσα το θεμητό ανταγωνισμό. Εκεί που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι βιοτέχνες, τα ελεύθερα επαγγέλματα δεν μπορούν να το κάνουν, το κάνουν οι μεγάλοι όμιλοι. Έπρεπε να δράσουμε και γι' αυτό αποτείω φόρο τιμή στον κύριο Κοφεράτη για την ποιότητα της δουλειάς του και για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξε και ο ίδιος αλλά και όλες οι πολιτικές ομάδες για να καταλήξουμε σε μια πρόταση ώστε να προστατεύσουμε τα δημόσια κατά των ε, εθνικών και ομιλικών συμφερόντων. Επίσης, ε, ε, ναι, κυρία Επίτροπε, όπως είπα, και στην τελευταία συνεδρίαση στον κύριο Μοσκοβισή ε, και στην ε, κυρία Τίσεν ε, στηριχτείτε, βασιστείτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αλλάξουν πια οι κανόνες λειτουργίας και η Ευρώπη να γίνει πιο διαφανής, πιο ανοιχτή, πιο ορατή και να πάψουν να υπερισχύουν τα προνόμια ορισμένων έναντι των δημόσιων συμφερόντων. Ευχαριστώ. Η κυρία Φεράρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Κοφεράτη για τη σκληρή και πολύ καλή δουλειά που έκανε. Το Κοινοβούλιο αύριο θα έχει τη δυνατότητα να εγκρίσει μια έκθεση που μπορεί να αποτελέσει καμπή στη διακυβέρνηση των εταιριών τόσο ως προς τη διοντολογία, αλλά και την πραγματική διαχείρισή τους. Εδώ χρειάζονται αυστηροί και κανόνες για την ε, διαχείριση των εταιριών, για τις αμοιβέ των διευθυντικών στελεχών και για τις πραγματικές επιδόσεις που πρέπει να συνδέονται με, την, ε, με τις αμοιβέ τους. Χρειάζεται η αρχή βάση της οποίας να αμείβεται η αφοσίωση του ε, διευθυντικού στελέχους, ο οποίος έχει την εταιρική ευθύνη και μπορεί να ασχολείται και με τα θέματα της κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που πρέπει να μας απασχολήσει είναι οι κανόνες που θα επιτρέπουν την, την ε, αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Οι, χώρες θα πρέ... οι εταιρείες θα πρέπει να πληρώνουν τους φόρους στις χώρες όπου βρίσκεται η έδρα τους. Και βεβαίως κυρίως θα πρέπει να ωφεληθούν οι πολίτες, διότι οι εταιρείες που περιβαλλοντικά και ηθικά είναι υπεύθυνε θα πρέπει να υπερασπίζονται το ευρωπαϊκό σύστημα ε, έναντι των κερδοσκόπων, που σήμερα εκμεταλλεύονται την κρίση από την οποία δυσκολεύεται να βρει διέξοδο σήμερα η Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπριουά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφοι, η χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε ότι τα τραπεζικά ιδρύματα ευνοούν τις, ε, τα βραχυπρόθεσμα εισοδήματα και πλήττουν το παραγωγικό μας μοντέλο. Οι επενδύσεις των ε, μετόχων πολλές φορές οδήγησε σε κίνδυνο τους επενδυτές και απειλήθηκε η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται στη διακυβέρνηση των εταιριών και ποιος είναι ο ρόλος των μετόχων και όλων των εμπλεκομένων. Η οδηγία αυτή ε, παροτρύνει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια μεταξύ των εταιριών στις σχέσεις τους και με τους επενδυτές. Εκτιμούμε ότι τα μέτρα που προτείνονται ε, οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως πιστεύουμε ότι τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να πάνε πιο μακριά, διότι θα πρέπει να είμαστε αφελείς αν πιστεύουμε ότι αυτό το εγχείρημα θα επιτρέψει το διεθνές χρηματοπιστωτικό ε, σύστημα να ελέγχεται καλύτερα. Είναι μεγάλη εμβέλεια οι προτάσει μα ε, για να φορολογήσουμε λόγω χάρη τι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ, την, να περιορίσουμε τη χρηματιστηριακή κερδοσκοπία και τα κέρδη των ε, μετόχων μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Φως. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε Επίτροπε. Στην Ευρώπη έχουμε ήδη ένα σύγχρονο εταιρικό δίκαιο που η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορεί να του προσθέσει πολλά. Κατά τη γνώμη μου όμως το θέμα της συμπερίληψης των εθνικών μετόχων στις εθνικές εταιρείες δεν ε, επιλύεται σωστά ούτε το θέμα των ε, ε, μειονοτήτων δηλαδή των μετόχων που έχουν λίγες μετοχές δεν ρυθμίζεται. Θέλαμε περισσότερα. Μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερα τις επιχειρήσεις. Δεν θα τις βοηθήσουμε όμως αν ενισχύουμε τα δικαιώματα των ε, μετόχων χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη συνολικότερα το θέμα λειτουργίας των επιχειρήσεων. Αυτό το σύστημα διαδικό, αυτό το διαδικό σύστημα με τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου και τα καθήκοντα του Εποπτικού Συμβουλίου εφόσον δεν υπάρχει και ένας σωστός ρόλος για την ε, ε, Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πρέπει να έχουν υποχρεώσεις και οι μέτοχοι. Θαυμάσια βέβαια είναι εργασία των σκιωδών εισηγητών και οδήγησε σε μια βελτίωση της συμβαστικής πρότασης και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μακροπρόθεσμα θα συμμετάσχουν περισσότερο οι μέτοχοι και στην δραστηριότητα των εταιριών και οι εθνικοί κανονισμοί δεν θα παραβιάζονται. Οι εκθέσεις αναχώρα είναι κάτι το οποίο δεν έπρεπε να μπει σε αυτήν την οδηγία διότι θα πρέπει να έχουμε διαφορετικού τύπου ρύθμιση σε διαφορετικά νομοθετήματα για τις εκθέσεις αναχώρα. Ο κύριος Χάουιτ. Ευχαριστώ, όπως και άλλοι. Καλωσορίζω την πρόταση για εκθέσεις αναχώρα, για να υπάρχει φορολογική ισότητα για όλους. Αλλά ως εισηγητής για την κοινωνική εταιρική ευθύνη, χαιρετίζω το ότι αναγνωρίζεται η ευθύνη των εταιριών, ότι αυτό είναι επίσης θέμα εταιρικής διακυβέρνησης. Πρέπει να έχουμε πιο μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση για να αντιμετωπίσουμε την κρίση και για να υπάρχει βιωσιμότητα. Η Επιτροπή έκανε μια ανακοίνωση που λέει ότι είναι υπέρ των μακροπροθέσμων επενδύσεων και το στηρίζω αυτό. Στηρίζω την οδηγία γιατί προσπαθεί να ενθαρρύνει την μακροπρόθεσμη προσέγγιση όπως ακριβώς προτείνει και το περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών καθώς και άλλες ε, δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών. Βεβαίως θα πρέπει να μπορούν να ψηφίζουν οι μέτοχοι για την αμοιβή των διοικητικών στελεχών και να ενημέρονται όλοι οι ε, εμπλεκόμενοι φορείς και όπως βλέπουμε πρέπει να αμείβονται όπως και σε άλλες περιστάσεις τα ηγετικά στελέχη όχι μόνο με την κερδοφορία αλλά και με βάση την βιωσιμότητα. Χαίρομαι που έχουν γίνει όλα αυτά αλλά δυστυχώς είναι λυπηρό ότι η δική μου κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι υπερβολική ρύθμιση αυτό που προτείνεται. Πρέπει οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν όλα τα θέματα που προκύπτουν τη δραστηριότητά τους και τα κοινωνικά και τα θέματα που είναι δικαιωματικά είναι σημαντικό ο νέος νόμος για τις εκθέσει για μη, δημοσιονομικά, για μη χρηματοπιστωτικά θέματα να ε, εφαρμοστεί. Ο κύριος Φόξ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Υποστηρίζω τη βελτίωση της ε, ε, συμμετοχής των μετόχων και την διαφάνεια, αλλά η έκθεση αυτή το παρακάνει, απομακρύνεται από αυτούς τους στόχους και σημαίνει περισσότερη άσκοπη γραφειοκρατία. Το άρθρο 3F, μπορεί να καταλήξουν στο να αποκαλύπτονται ευαίσθητε εμπορικά πληροφορίε χωρίς να ωφελεί το κοινό. Γιατί κάποιο ο οποίο δεν χειρίζεται ενεργητικά να είναι απεύθυνο για να μειώνονται οι ε, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ε, ε, ευθύνες συγγνώμη, να μειώνεται η έκθεση σε τέτοιου κινδύνου αυτός στου οποίου επενδύει. Και δεν συμφωνώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εισάγουν επιπλέον μέτρα για να υποστηρίξουν τη μακροπρόθεσμη επένδυση. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν την ευθύνη. Και αυτό που παίζει ρόλο είναι να είναι μακροπρόθεσμες οι επενδύσεις και όχι μακροπρόθεσμη κατοχή των ε, μετόχων. Το να συμπεριλάβουμε επίσης ε, την υποβολή εκθέσεων αναχώρα για όλες τις μεγάλες εταιρείες δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει τα δικαιώματα των μετόχων. Και είναι απαράδεκτο αυτή από την αριστερά του σώματος να συμπεριλαμβάνουν τέτοιες υποχρεώσεις σε διάφορα θέματα. Αντίθετα πρέπει να προωθήσουμε αυτά που κάνει ο ΣΑΚ και το G20 σε διεθνές επίπεδο του θέματος αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μποργέτσιο. Πρόεδρε, η αφοσίωση της ηγετή, όμως η Ευρώπη ακόμη δεν έχει πραγματοποιήσει μια αληθινή οικονομική δημοκρατία ιδίως για τις εταιρικές υποχρεώσεις και την προσώπηση των μικρών μετόχων ιδίω κατά ένα τρίτο στο Διοικητικό Συμβούλιο των Εταιριών. Από αυτή τη σκοπιά, γιατί δεν σκεφτόμαστε να οργανώσουμε εκλογέ για να υπάρχει άμεση εκπροσώπηση των νόμιμων συμφερόντων των μικρότερων μετόχων, οι οποίοι πολλέ φορέ εκπροσωπούν το εργατικό δυναμικό, τους εργαζομένους. Εκεί θα πρέπει να δώσουμε ε, προσοχή στις μεγαλύτερες εξουσίες. Και επίσης να επιβληθούν κυρώσεις στις εταιρείε όπου οι διευθυντές τους το ε, παρεμποδίζουν αυτό ε, όταν δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια για τον ε, κύκλο εργασιών, τον ισολογισμό των εταιρεών και τις πληροφορίες, θα πρέπει να, να λαμβάνουμε υπόψη και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης, θα πρέπει, εφόσον αυτό το σύστημα ολοκληρωθεί και υλοποιηθεί, να επιτρέψει να υπάρχει εμπιστοσύνη από την πλευρά των πολιτών για τις πληροφορίες που δίνονται και προς τους θεσμικούς φορείς. Πρέπει να περιοριστεί αυτή η αδιαφάνεια που βαραίνει την δραστηριότητα κυρίως των μεγάλων πολυεθνικών αλλά και όλων των επιχειρήσεων. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπέκερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλωσορίζω αυτήν τη σημαντική έκθεση. Καθορίζω αυτός, ε, καλωσορίζω αυτούς τους ε, σημαντικούς στόχους για την μακροπρόθεσμη συμμετοχή των μετόχων. Είναι θετικές αυτές οι εξελίξεις από την προηγούμενη Ολομέλεια. Έχει βελτιωθεί το νομικό κείμενο και με ενδιαφέρει πάρα πολύ και ως Αυστριακός. Η παραδοσιακά επιτυχής δομή Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου να διατηρηθεί και να μην υπάρξει μεταφορά αρμοδιοτήτων. Όμως φαίνεται ότι είμαστε εξαίρεση. Είναι όμως περίεργο το ότι διαπιστώσαμε ότι και μεταξύ των σοσιαλιστών εδώ στο σώμα έγιναν προσπάθειες ούτω ώστε τα εποπτικά συμβούλια που για μας είναι δεσμευτικά και είναι δεσμευτικό να συμμετέχουν τα δικαιώματα των εργαζομένων να αποφασίζουν τα εποπτικά συμβούλια γίνεται προσπάθεια και για το δικαίωμα των αμοιβών των ηγετικών στελεχών. Δεν είναι δυνατόν το εποπτικό συμβούλιο να έχει για τα θέματα αυτά περισσότερες αρμοδιότητες από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επίσης, ο καθορισμός των μετόχων και η δυνατότητα δημοσίευσης των ονομάτων τους πρέπει να βασιστεί στις ε, παραδοσιακές ε, λειτουργίες των επιχειρήσεων. Δεν θα πρέπει βέβαια όλα αυτά να οδηγήσουν σε εθνικιστικές και εθνικές γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις. Περιμένουμε λοιπόν από τον ε, τριμερή διάλογο να ληφθούν υπόψη αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στάινμπρουκ. Η κυρία Στάινμπρουκ. Ο Σέτζο Κομφεράτη βελτίωσε κατά πολύ την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση που έχουμε τώρα ενώπιον μα ενισχύει τη διαφάνεια τη ε, λειτουργία των επιχειρήσεων. Όμω δυστυχώ το κείμενο αυτό δεν ε, εμπλέκει αρκετά του εργαζομένου στη λήψη αποφάσεων. Ερωτώ του συνδημοκράτε και φιλελεύθερου συναδέλφου, την πλειοψηφία του, γιατί αντιτίθεστε τόσο πολύ κατά τη συμμετοχή των εργαζομένων. Μα οι εργαζόμενοι έχουν κάθε συμφέρον στο να επιτύχει μια επιχείρηση, να έχει μακροπρόθεσμο μέλλον. Επίσης λυπηρό είναι ότι η Γενική Συνέλευση των εισηγμένων εταιριών κάθε τρία χρόνια θα αποφασίζει δεσμευτικά για τις ε, αμοιβέ. Δεν υπάρχει ισορροπία λοιπόν μεταξύ των διαφορών πλευρών. Οι μέτοχοι θα έχουν πολύ μεγάλο ειδικό βάρος και μερικοί μέτοχοι με ε, ε, ιδιαίτερα συμφέροντα θα μπορέσουν να παίξουν πολύ αρνητικό ρόλο. Η κυρία Φανστόρχ, έχει, υπάρχει γαλιάζω και κάρτα για σας. Τη δέχεστε? Όχι. Δεν θέλει να απαντήσει η συνάδελφος. Η κυρία Φανστόρχ. Yeah, Σήμερα συζητάμε για το φορολογικό απόρριτο των επιχειρήσεων. Και όλοι κάθε είδους αριστεροί θέλουν να το καταργήσουν. Να τότε να το κάνουμε για όλους. Ο καθένας να ξέρει ποιος πληρώνει πόσους φόρους σε κάθε χώρα. Αυτό θα ήταν ε, διαφάνεια για όλους. Όμως οι επιχειρήσεις ε, δεν είναι υπόλογες έναντι του κάθε πολίτη. Είναι υπόλογοι έναντι των μετόχων και έναντι της εφορίας. Εσείς λέτε ότι ε, θα ρίξετε φως στο σκοτάδι. Αντίθετα, εγώ νομίζω ότι παραβιάζονται απόρριτα. Στη Φινλανδία, μια φορά το χρόνο, ε, δημοσιεύεται ποια είναι τα κέρδη μιας επιχείρησης και πόσα πληρώνει ως ε, εταιρεία στην εφορία. Και ορισμένοι το αποκαλούν αυτό δημοσίευση της ζήλιας. Ορισμένοι θα ζητήσουν και από τους πολίτες, αν το ζήτησουμε από τις αυτό μετά, να μας λένε πόσα πληρώνουν. Τα απορρίπτω και τα δύο. Ο κύριος Μπρετό. Ο κύριος Λεμπρετών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το κείμενο αυτό σκοπό έχει να αντικαταστήσει τον οικονομικό καπιταλισμό με έναν υπεύθυνο καπιταλισμό. Στόχο του είναι να παροτρύνει του επενδυτέ να διατηρήσουν τι μετοχέ του για πιο πολύ καιρό και να μην έχουν τον πειρασμό να κάνουν ε, κέρδο βραχυπρόθεσμα. Το κείμενο προσπαθεί να εντοπίσει του μετόχου. Ε, άλλο εντοπισμό καλώ ακούγεται, όμω θα πρέπει στην, ε, στο καταστατικό τη κάθε εταιρεία να έχει ένα κατάλογο των μετόχων, των μετόχων για σκοπού διαφάνεια. Θα πρέπει Όμω όμως να μην επιφέρει και υπερβολικό κόστος μια τέτοια ε, καταλογοποίηση. Θα πρέπει λοιπόν οι μέτοχοι που κρατούν τις μετοχές τους για πάνω από δύο χρόνια να έχουν δικαίωμα διπλής ψήφου. Αυτό το δικαίωμα της διπλής ψήφου είναι μια καλή ιδέα εάν οι δικαιούχοι είναι τα κράτη μισθωτή της επιχείρησης. Διότι τότε θα μπορέσουν να ε, αποφύγουν την ανάληψη του ελέγχου από ξένες επιχειρήσεις. Έτσι η διπλή ψήφος θα είναι ένα εργαλείο πατριωτισμού, οικονομικού πατριωτισμού. Ευχαριστούμε κύριο Σβάμπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν στην εξέβρεση συμβασμού. Γιατί καταφέραμε λοιπόν να έχουμε μια κοινή γραμμή. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Ταντέο Σίφκα Σκιώδη και τον Σέρζο Κομφεράτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πεπισμένος ότι ο στόχος για μια βιώσιμη ανάπτυξη της ε, μιας εταιρείας και ο στόχος μιας διαφάνειας, όλα αυτά μας συνδέουν. Σε όλα αυτά συμφωνούμε. Το ερώτημα μόνο είναι ε, σε τι βαθμό τα επιτυγχάνει αυτή η οδηγία αυτά. Και πολλοί λένε ότι το βασικό είναι οι εκθέσεις αναχώρα. Τώρα δεν είμαι η για τέτοια θέματα λογιστικά, αλλά στην τάξη την προηγούμενη εβδομάδα Ακούσαμε έναν καθηγητή για φορολογικά θέματα που μας είπε ότι και με τις εκθέσεις αυτές... Α, ήταν Βρετανός, ήταν Βρετανός, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι ε, είναι ευρέως διαδομένες αυτές οι ότι οι εκθέσεις αυτές στο τέλος δεν θα βλέπουμε τις μεταφορές στο εσωτερικό των εταιριών. Και το πρόβλημα με τους μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους δεν είναι διαφάνεια αναχώρα, αλλά το ότι δεν ξέρουμε πώς είναι οι χρηματοδοτικές και χρηματοπιστωτικές δομές μέσω των, και μεταφορές μέσω των, ε, στο εσωτερικό των εταιριών, μέσω για παράδειγμα των διπλωμάτων βρεστεχνίας κτλ. Το πρώτο βήμα ωστόσο ε, γίνεται με αυτό το κείμενο. Το δεύτερο, όπως είπε και ο Σνάλφος Μπέκερ, αφορά το ότι πρέπει να βρούμε λύσεις που να μπορούν να λειτουργήσουν σε όλες τις χώρες μέλη και υπάρχουν διάφορα και διαφορετικά πρότυπα στο εταιρικό δίκαιο των διαφόρων κρατών μελών. Νομίζω όμω ότι μέσω των τροπολογιών οι συμβασμοί είναι καλοί. Και παρακαλώ τον εισηγητή από κοινού να εξετάσουμε περαιτέρω δυνατότητε, ούτω ώστε στο τέλο να επιτύχουμε τον κοινό μας, στόχο. Ακόμη απέχει, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να τον επιτύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σφάμπ, υπάρχει μια μπλε κάρτα, τη δέχεστε. Ο κύριο Φρουντζούλικα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Σφάμπ, είπατε, για να έχουμε μακροπρόθεσμες επενδύσεις, για να ενισχύσουμε αυτές τις επενδύσεις, είπατε κάτι. Κύριε Σφάμπ, για να προωθήσουμε τη διατήρηση μετοχών για μεγάλο χρονικό διάστημα, μάλλον να κάνω την ερώτηση, Εάν υπάρχουν, υπάρχει μακροπρόθεσμη κατοχή μετοχών, σημαίνει ότι υπάρχουν και μακροπρόθεσμε επενδύσει. Μήπω δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την ερώτησή σα. Εγώ πιστεύω ότι μπορώ να πω ότι όποιο θέλει να προωθήσει το ενδιαφέρον κάποιων επενδυτών και ιδιαίτερα όσον αφορά τα μπόνου, είναι σημαντικό να διατηρούνται οι μετοχέ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τι περαιτέρω βήματα μπορούμε να κάνουμε Μπορούμε να το δούμε. Είμαι βέβαιος ότι στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου θα το συζητήσουμε. Και δεν τα ξέρω λοιπόν σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τζιλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι είναι, η έκθεση αυτή είναι σημαντικό βήμα, όχι για την αντιμετώπιση του θέματος της άσκησης δικαιωμάτων των μετόχων, αλλά και της πάταξης της φοροδιαφυγής. Και είναι ένα από τα πρώτα θέματα στο πλαίσιο της συνομοθεσίας ε, που έχουμε λόγο κοινοβούλια για φορολογικά ζητήματα. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ε, σε ό,τι αφορά τους φόρους που καταβάλουν οι εταιρείε. Αν ακολουθούν όμως τους κανόνες, ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα. Υπήρξαν ε, διάφοροι ειδικοί που λένε ότι οι χώρα είναι ένας τρόπος ε, να έχουμε αποτελέσματα και προτεραιότητα για τη δική μου ομάδα είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής. Αυτό το οποίο λοιπόν είναι κρίσιμο για τους ε, μεγαλομετόχους είναι να συνεχίσουν να αφισβητούν ή να θέτουν τέλο πάντων τις πολιτικές ε, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η δεξιά μελων του διοικητικου συμβουλιου δεξια μιλα και αυτή για τη φοροδιαφυγή. Αλλά ας είμαστε σοβαροί. Θα πρέπει να γίνουν τα λόγια πράξη όλοι θέλουμε την διαφάνεια για τα φορολογικά ζητήματα, ιδίως γιατί οι ίδιοι οι απλοί πολίτες κάνουν φορολογικέ δηλώσει, δέχονται περικοπές στι υπηρεσίες, ενώ οι πολυεθνικές ξεφεύγουν και πληρώνουν πολύ λίγους φόρους ακόμη. Ξέρω ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων έλαβε μια ξεκάθαρη δημοκρατική απόφαση και ελπίζω το Κοινοβούλιο να μεταλλευτεί την ευκαιρία και αύριο να ψηφίσει θετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ με τέσσερα μου να συγχαρώ όσους εργάστηκαν για την έκθεση αυτή. Είναι μια καλή αρχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να θέσει ως στόχο την διαφύλαξη των φυστάμενων θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων. Πρέπει επίσης να αυξήσει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά. Θέλουμε μια εναρμονισμένη νέα προσέγγιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι αναγκαίο να υπάρξουν τα ε, ενιαία πρότυπα για όσες εταιρείες ε, εργάζονται μακροπρόθεσμα προς το συμφέρον και των εταιρεών και των κρατών μελών εν γέννη. Επίσης, θα πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφενός, της εγγύησης ε, και της εγγύησης των δικαιωμάτων των μετόχων, αλλά και της διατήρησης ενός ε, παρκούς επίπεδου διαφάνειας αφετέρου. Χαιρετίζω το γεγονός ότι υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. και οι εταιρείε είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να καταρτίζουν ε, τα σχέδιά τους σε ό,τι αφορά και τις αποδοχές των ε, δικτικών ε, στελεχών. Ωστόσο, η εταιρική διακυβέρνηση είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει και τους εργαζομένους. Η δηλαδή, συμμετοχή των εργαζομένων είναι σημαντική. Ο κύριος Νεγκρέσκου. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ τον εισηγητή για τις προσπάθειές του και για την ε, σύνταξη της έκθεσης αυτής που είναι σαφέστατη και περιλαμβάνει τις βασικές προτεραιότητες που συζητήθηκαν και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Ο ρόλος των εργαζομένων, των μισθωτών, των θεσμικών επενδυτών και γενικώ των μετόχων στην ιατρική διακυβέρνηση βρισκόνται στην καρδιά του κειμένου το ίδιο και οι αμοιβέ και το φορολογικό σύστημα στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό για τους πολίτες και την ε, Ευρώπη να γνωρίζουν πόσους φόρους πληρώνουν οι πολυεθνικές εταιρείες. Πρέπει να είμαστε σε θέση να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή και εδώ στο Κοινοβούλιο να προτείνουμε μια λύση που να μας επιτρέψει να αποφύγουμε την επανάληψη καταστάσεων όπως το LuxLeaks στο μέλλον. Ευχαριστούμε. Επόμενος συνάδελφος για μισό λεπτό, ο κύριος Μπέντσιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σημαντική η συμβολή των μετόχων στην ε, εταιρική διακυβέρνηση και βεβαίως ως μέτοχος κανείς πρέπει να λαμβάνει μέρος στην διαδικασία λήψη αποφάσεων. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όμως πηγαίνει αρκετά μακριά. Θα δημιουργεί το ένα σύστημα πολύ αδιάλακτο πολύ αυστηρό που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εθνικές επιλογές σε ό,τι τη ρύθμιση της δράσης των μετόχων. Θα πρέπει να αποφύγουμε την ε, ανάκαμψη της ε, πορείας των επιχειρήσεων προς την ανάπτυξη. Στη συμβαστική λύση του Κοινοβουλίου νομίζω έχουμε μία λύση που επιτρέπει να περάσουμε σε ενδιαφέρουσες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαπάτης είναι σημαντικά στοιχεία επίσης και συνεργαζόμαστε με τις ε, αρμόδιες αρχές για το σκοπό αυτό. Θα πρέπει σε αυτή την οδηγία να διατηρήσουμε αμύωτη αυτή την πορεία για να ρυθμίσουμε όχι τη δράση των επιχειρήσεων αλλά των μετόχων. Θα πρέπει και η φορολογική μας νομοθεσία να συμπλέψει και να καταφέρουμε να έχουμε αποτελεσματική δράση για τους μετόχους. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό κύριο κύριος Με συγχωρείτε, γαλάζια κάρτα. Δέχεστε γαλάζια κάρτα. Κύριε Μπέντσεν. Έχετε 30 δευτερόλεπτα. Όχι 30 λεπτά. Ζέστητε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Μπένσον δεν θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει δίκαιο και θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ των ε, εταιριών και με την ε, αναχώρα υποβολή εκθέσεων. Να υπάρχει ένα αυξημένο επίπεδο διαφάνεια για να αποφύγουμε τι φοροαπάτε και φοροδιαφυγέ τέτοια φαινόμενα δεν είναι σημαντικό το σύστημα από πολλές εκθέσεων ανά χώρα. Θα μας στηρίξετε κυρία Μπέντσεν σε αυτό το reporting και τις σχετικές προτάσεις. κοιτάξτε, νομίζω ότι αρκεί να έχουμε γενικού κανόνες διαφάνειας. Ναι, ας έχουμε υποβολή εκθέσεων χώρα, αλλά στην ε, προκειμένη περίπτωση έτσι κι αλλιώ μιλάμε για μια οδηγία και το δίκαιο θα διέπει ε, τη δράση των ε, ε, μετόχων. Όχι την φορολογική νομοθεσία. Δεν θα συμπεριλάβουμε όλε τι πρωτοβουλίε εδώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάγκη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Όπως είδαμε μέσω των LuxLeaks, Υπάρχει πρόβλημα έλλειψης ε, διαφάνειας. Και αυτό που χρειαζόμαστε είναι να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή. Τα σκάνδαλα του LuxLeaks ε, μας βοήθησαν να καταλάβουμε τι χρειάζεται να κάνουμε. Χρειαζόμαστε περισσότερη πληροφόρηση. Γιατί αλλιώ, αν δεν περιέχει πληροφορίε, η διαφάνεια δεν σημαίνει τίποτα. Η υποβολή εκθέσεων αναχώρα είναι ζωτική για να έχουμε αυτή την αναγκαία πληροφόρηση. Πρέπει να υπάρχουν βεβαίω αμοιβέ για τα διοικητικά στελέχη, αλλά πρέπει να είναι λογικέ, δίκαιε αυτέ οι αμοιβέ. Και αν δεν έχουμε πληροφόρηση γι' αυτό, τότε δεν μπορούμε φυσικά να το ελέγξουμε. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν εκθέσει από αυτού. Αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε και περισσότερα. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους κοιόδης γιατί επέτυχαν ήδη σημαντική πρόοδο να αφορά την ασφάλεια. Την διαφάνεια, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητή για ένα λεπτό ο κύριος Πυρίνσκι. Ευχαριστώ. Το βασικό θέμα πιστεύω της έκθεσης αυτής που θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι είναι ότι δίνει κάθε κίνητρο για υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση όλα τα μέτρα που αναφέρονται στα δικαιώματα των μετόχων και άλλων εμπλεκομένων, η ανάγκη για σαφείς εκθέσεις και για τις αμοιβέ, αλλά και για το κόστος και τα κέρδη, οι εκθέσει αναχώρα, όλα αυτά είναι πολύ σωστά προσανατολισμένα, ούτω ώστε να έχουμε ένα νέο επίπεδο ποιότητας εταιρικής διακυβέρνησης που θα αναπροσανατολίσει την συμπεριφορά πέρα από την βράχυπρόθεσμη αντιμετώπιση για έναν υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας για να εξυπηρετήσουν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων, των ε, εμπλεκομένων και της κοινωνίας. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό, λέει η πρόεδρος τώρα. Αν δεν κάνω λάθος. Α, όχι, ένα λεπτό. Η κυρία Γοζιέρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, με μία λέξη μπορούμε να χαιρετήσουμε αυτή την έκθεση. Μπράβο, μπράβο στον Σέρτζο Κοφεράτη για την αξιοσημείωτη δουλειά που έκανε σε σχέση με την οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων. Ε, σημαντική πρόοδο με το κείμενο αυτό για να ενισχύσουμε τι μακροπρόθεσμε επενδύσει και τη διαφάνεια διαχείριση των επενδύσεων. Έχουμε μείζονη, μείζονο πρόοδο. Επιτέλου ε, θα μπορέσουμε με τι εκθέσει αναχώρα να εντοπίζουμε του χειρισμού ε, επιθετικού φορολογικού ε, σχεδιασμού οι πολυεθνικές θα πρέπει να πληρώνουν εκεί που ε, παράγουν κέρδος και στους ε, φορολογικούς παραδείσους ώστε να μπορούν να βλέπουν οι πολίτες και οι αρχές που πηγαίνουν οι φόροι. Παρά την προσπάθεια των συναδέλφων της δεξιάς να καταργήσει τα μέτρα διαφάνειας, δεν το πέτυχαν. Αν θέλουμε να μην επαναληφθεί το σκάνδαλο LuxLeaks και να στηρίξουμε τις ΜΜΕ που δημιουργούν θέσεις εργασίας ε, που και πληρώνουν φόρους και αν θέλουμε να αποφύγουμε τη φοροαποφυγή από τις μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να στηρίξουμε αυτά τα μέτρα διαφάνειας. Ελπίζω αύριο να υπάρξει μεγάλη πλειοψηφία για τη στήριξη των μέτρων που εμείς έχουμε προτείνει ως σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ελπίζουμε να δείξει ότι ανταποκρίνεται τις προσδοκίες των συμπολιτών μας ε, το κοινοβούλιο διακόπτεται. Είχατε μόνο ένα λεπτό, λυπούμε, λέει πρόεδρο. Θα πάμε στον επόμενο ομιλητή που και αυτό έχει ένα λεπτό στη διάθεσή, τον κύριο Κόφοντ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπη, Φυσικά και είναι σημαντικό να υπάρχει ένα κράτος ε, πρόνοιας. Βέβαια ε, όλα αυτά κοστίζουν, κοστίζουν χρήματα και είναι τα χρήματα που πληρώνουμε με τους φόρους. Πολλές φορές όμως ε, οι μεγάλες επιχειρήσεις πολύ εύκολα ε, καταφεύγουν σε πρακτικές ε, φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής. Ε, είναι ένα είδος αθλήματος για μεγάλες επιχειρήσεις θα έλεγα. Επίσης άλλες επιχειρήσεις προβαίνουν σε παρακινδυνευμένες επενδύσεις με υψηλές αποδόσεις και όλα αυτά οδήγησαν και ολόκληρες χώρες στην κρίση. Θα πρέπει να στηρίξουμε την ανάπτυξη και τις αξίες μας με αυτή την ε, οδηγία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ε, τις ανεύθυνες αυτές ε, επενδυτικές πρακτικές. Θα πρέπει λοιπόν και εκθέσει αναχώρα να χρησιμοποιηθούν για να μπορούμε να βλέπουμε ποιες είναι οι χρηματοοικονομικές ροές και να πληρώνουν οι επιχειρήσεις εκεί που κερδίζουν τα χρήματά τους. Και βέβαια να αποφύγουμε και τους φορολογικούς παραδείσους. Ευχαριστώ πολύ. Γκόμες. Μπράβο στον ε, Σέρτζο, μπράβο στην Επιτροπή Γιούρη και μπράβο στο Κοινοβούλιο για την έκθεση αυτή κοφεράτη που θα ενισχύσει την ε, διαχείριση των φορολογικών ε, συστημάτων με πληροφορίες για τους δημοσιογράφους και τους πολίτες ώστε να μην υπάρχει φοροδιαφυγή, φοροαπάτη, κατάχρηση και η διαφθορά που όλα αυτά επιτρέπουν να σοβεί. Η ε, περίπτωση του Swissleaks και του LuxLeaks δείχνουν στην Ευρώπη πόσο αυτά τα σκάνδαλα πλήττουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα αλλά και σε άλλες χώρες αναπτυσσόμενες. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα ε, για το οποίο δεν μπορούμε να αφήσουμε τις φορολογικές διοικήσεις να λάβουν μόνο τις αποφάσεις, γιατί δεν έχουν πάντοτε τους πόρους και τις επενδύσεις που χρειάζονται ή με τις πολιτικές λιτότητας περιορίζονται και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πολυεθνικές που ουσιαστικά υπερβαίνουν την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτή η έκθεση λοιπόν με την υποβολή εκθέσεων αναχώρα επιτρέπει υποχρεωτικά να διευρυνθεί το σύστημα της διαφάνειας σε όλες τις πολυεθνικές επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς δράσης τους. Ευχαριστούμε και για ένα λεπτό η κυρία Ντότζ. Ευχαριστώ. Πολλά στοιχεία της έκθεσης αυτής είναι θετικά. Αλλά θέλω να μιλήσω για τα θέματα εκθέσεων αναχώρα. Όπως υπόθηκε, αυτό θα σήμαινε ότι οι πολυεθνικές θα πρέπει να αναφέρουν πως είναι οι εργαζόμενοι της, ποιος είναι ο κύκλος εργασιών και τους φόρους πληρώνουν σε όλες τις χώρες της Ένωσης όπου δραστηριοποιούνται. Αυτές οι εκθέσεις πρέπει να είναι δημόσιες. Πρώτον γιατί έτσι οι μέτοχοι και οι επενδυτές χρειάζονται αυτή την πληροφόρηση για να κάνουν τις, ε, πάρουν τις αποφάσεις τους. Δεύτερον, γιατί είναι δικαίωμά μα ω πολίτε και ω καταναλωτέ να έχουμε αυτή τη βασική πληροφόρηση για τη λειτουργία των εταιριών που λειτουργούν στι χώρε μα. Τρίτον, διότι οι περισσότερε επιχειρήσει ήδη χορηγούν αυτή την πληροφόρηση γιατί βασίζονται μόνο σε μία χώρα. Και χρειαζόμαστε αυτή την προφόρηση, ούτω ώστε οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, οι δημοσιογράφοι, οι πανεπιστημιακοί, καθώ και οι εφορεί να μπορούν να δουν πού υπάρχουν ενδεχόμενα καταχρήσεων. Α αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να βελτιώσουμε την κατάσταση και για του μετόχου και για του άλλου επενδυτέ και πρώτα απ' όλα για του φορολογούμενου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρο. Ε, τώρα, επειδή έχουμε πολλού για τη διαδικασία προσέλκυση τη προσοχή, σα παρακαλώ, εάν βοηθήσετε και διατηρήσετε το χρόνο σα, θα μπορέσουν όλοι να πάρουν το λόγο. Δίνω λοιπόν το λόγο στην κυρία Σούλιαν. Ευχαριστώ πολύ. Υποστηρίζω την ε, τροποποίηση της οδηγίας ούτως ώστε να ε, εμπλέκονται μακροπρόθεσμα οι επενδυτές. Το θέμα είναι οι επιχειρήσεις να δημοσιοποιούν τις ε, πληροφορίες στις χώρες όπου φορολογούνται. Οι μικρομεσαίες ε, είναι σε θέση έναντι των πολυεθνικών που ε, μεταφέρουν τα κέρδη τους σε φορολογικούς παραδείσους. Εάν οι επιχειρήσεις ε, δημοσιοποιήσουν περισσότερα στοιχεία, θα οδηγήσει αυτό και σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Γιατί όλοι θα έχουν τα στοιχεία υπόψη τους και θα γνωρίζουμε πού είναι ασφαλείς οι επενδύσεις. Οι πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη ή που θα θέλουν να δραστηριοποιηθούν αξιοποιούν τη δυνατότητα φορολογικού ανταγωνισμού. Γι' αυτό είναι αναγκαία η διαφάνεια που θα επιτευχθεί μέσω της ε, τροποποίησης της οδηγίας. Έτσι λοιπόν θα βοηθήσουμε τους επενδυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ πρόεδρε στην παρέμβασή μου μίλησα για τις αρχές της διαφάνειας, της αφηνής και της ε, πληροφορία ενημέρωσης για κάθε είδους οικονομικό στοιχείο. Εδώ μπορούμε να καλλιεργήσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού και να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για την κατάσταση των μετόχων και την εταιρική διακυβέρνηση. Με εμπιστοσύνη στο νομισματικό και οικονομικό σύστημα και το τι συμβαίνει στο τραπεζικό σύστημα. Έτσι, οι πληροφορίε μπορούν να διασυνδεθούν με το επίπεδο συμμετοχή και την εταιρική διακυβέρνηση. Οι μέτοχοι θα πρέπει να μπορούν ανάλογα με τι επενδύσει του και για τις εισηγμένε χρηματιστηριακέ εταιρείε, να υπάρχουν απαραίτητε ε, πληροφορίες για τους φορείς και τις ε, φορολογικέ αρχές. Μπορούμε έτσι να δούμε τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα των ε, εταιριών και να βλέπουμε ποια είναι τα χρηματοπιστωτικά και μη ε, αποτελέσματα μιας εταιρείας. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής, κυρία Τόμαφιτς. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σωστά αναγνωρίζει ο εισηγητή την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια ε, στι εισηγμένε στο χρηματιστήριο εταιρείε. Δεν είμαι βεβαία κατά πόσον όμω ο στόχο αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τι προτινόμενε στην έκθεση μεθόδου, ε, ιδίω ε, με τη συσσόρευση απαιτήσεων για συγκέντρωση στοιχείων ε, και υποβολή εκθέσεων κτλ. κτλ. Επίσης, η συμμετοχή των μετόχων ε, στα θέματα που αφορούν τη διαχείριση των εταιρεών είναι κάτι ευκταίο. Όμως, η ε, ανταλλαγή πληροφοριών για την ταυτότητα όλων των μετόχων σε έναν μέτοχο δεν ξέρω κατά πόσον θα ήταν εφικτό αν δεν προηγεί το η συγκατάθεση όλων των άλλων μετόχων. Επίσης μπορεί αυτό να αυξήσει τη γραφειοκρατία. Για το γραφειοκρατικό άκτος καλό είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον σταθερό που θα ε, ε, φέρει περισσότερη πρόβλεψιμότητα και θα βοηθήσει την υπόθεση των αγορών επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό. Ο κύριος Γιακόβιτ. Ευχαριστώ πολύ. Αναφίβολα η συζήτηση αυτή και το γεγονό ε, ότι έχει προκληθεί παρόλα αυτά κρίση σημαίνει ότι χρειαζόμαστε τροποποίηση της νομοθεσίας για τις εταιρείες, τη διακυβέρνησή τους και τους μετόχους. Συμφωνώ λοιπόν με αυτήν την έκθεση λόγω των και των συμβαστικών συμβιβασμών οι οποίοι επετέφθησαν γιατί πρέπει να μπορούμε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι μέτοχοι όλων των εισηγμένων εταιρεών. Χρειαζόμαστε διαφάνεια. Γιατί αυτό θα εγγυηθεί μια πολύ καλύτερη κατάσταση για τις δυνατότητες καταπολέμησης ε, της ε, φοροδιαφυγής και όλα τα άλλα όσα έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Και οι εκθέσει αναχώρα είναι χρήσιμε. Είμαι πεπισμένο γιατί είναι διαφορετική η κατάσταση από χώρα σε χώρα. Και γι' αυτό θα επιτύχουμε συνεργείες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η οδηγία σκοπό έχει να στη λύση αποφάσεων των επιχειρήσεων. Και το ίδιο και για τις επιχειρήσεις που, ε, έχουν, που ασχολούνται με τα βραχυπρόθεσμα ωφέλη τους και ουσιαστικά ε, διακυβεύεται έτσι η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ίδιας της εταιρείας δεν πρέπει να αγνοούμε, είναι υπογνώμαστε ότι αγνοούμε ότι και η μετοχή που επιδιώκουν πρόθεσμα ωφέλη, όπως το κείμενο ορίζεται μεταξύ ε, του ε, μέσου και του βραχυπρόθεσμου ε, μετόχου, θα πρέπει παρόλα αυτά να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή των μετόχων και τις επενδύσεις που γίνονται. Η οδηγία θέτει βεβαίως την αντίστροφη ερώτηση, δηλαδή η λύση για τη λήψη αποφάσεων στις εταιρείε για να είναι βιώσιμη και ε, μακροπρόθεσμη θα πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική διαφάνεια και την, ε, ήδη, την συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων και τους τοπικούς ε, συμμετέχοντες στην όλη διαδικασία και διακυβέρνηση της εταιρεία. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σόλτερς. Πριν από 15 χρόνια, τέτοιες προτάσεις θα είχαν αντιμετωπίσει πολύ σοβαρή αντίσταση. Σήμερα βέβαια έχει αλλάξει η κατάσταση. Διότι ε, έχουμε περάσει από μια πολύ ε, οδυνηρή χρηματοπιστωτική κρίση και έχουμε και το θέμα των LuxLeaks και όλοι ξέρουμε πώς λειτουργούν οι φορολογικοί παράδεισοι. Όλα αυτά έπεισαν την κοινή γνώμη ότι χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια για τον τρόπο λειτουργίας ε, και διοίκησης των επιχειρήσεων. Και αυτό ισχύει κυρίως για τις πολυεθνικές. Πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια. Τώρα για τις εκθέσεις αναχώρα. Πρέπει οπωσδήποτε και αυτές να υπάρχουν για να υπάρχει περισσότερη εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις. Εάν επιτύχουμε αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε στο μέλλον μπορούμε να ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχουν εταιρείε που θα παραβαίνουν του κανόνε. Ελπίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη τη επιχειρήση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η έκθεση που έχουμε ενώπιόν μα προσπαθεί να συμμετέχουν περισσότερο οι, μετοχοί στον τρόπο, οι μέτοχοι στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και τον καθορισμό των αμοιβών και την διακυβέρνηση. Και προβλέπονται περισσότερες δυνατότητες γενικά για τους μετόχους. Ε, ένα τμήμα του νόμου Φλωράνς της προηγούμενης, ε, της περσινής χρονιάς είναι ε, οπωσδήποτε πρόδρομος αυτής της σημερινής νομοθεσίας. Όμως στη Γαλλία υπάρχουν πολλές επικρίσεις και από τον Bloomberg υπάρχουν επικρίσεις για αυτό το νόμο γιατί λέγεται ότι ορισμένοι κύριοι μέτοχοι που στη Γαλλία είναι το κράτος, έχουν διπλό δικαίωμα ψήφου και είναι σε μειονεκτική θέση οι μικρομέτοχοι. Στην ουσία δηλαδή ευνοούνται οι θεσμικοί επενδυτές. Υπάρχουν λοιπόν θετικά, αλλά υπάρχουν και αρνητικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριο Σκέλη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι πηγαίνει προς την κατεύθυνση η έκθεση αυτή, ωστόσο δεν έχουμε ακόμη επιτύχει το στόχο μας. Για παράδειγμα, ορισμένα από τα θετικά σημεία είναι ότι θα δοθεί μεγαλύτερη σημασία στις επενδύσεις σε εταιρείε. Πολλές φορές γίνονται επενδύσεις, αλλά καταλείπεται η εταιρεία στη συνέχεια. Είναι λοιπόν σημαντικό ε, να στηριχθεί, να εξακολουθήσει να στηρίζεται εν λόγω εταιρεία. Επίσης καλό είναι να πιέσουμε τις εταιρείε ώστε να πληρώνουν ε, το μερίδιο των φόρων που τους αναλογεί και να τυπώνονται οι σχετικές συστάσεις αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα σχόλια που ακούστηκαν νωρίτερα, ότι δηλαδή εκθέσει αναχώρα δεν είναι επαρκή ρύθμιση ε, για την επίτευξη αυτών των στόχων. Νομίζω λοιπόν ότι η Κομισιόν θα πρέπει να ακούσει τι φωνέ των Ευρωβουλευτών και να λάβει σοβαρά υπόψη τις απόψεις Μα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Φρουντζουλίτσα δεν νομίζω ότι είναι στην αίθουσα, οπότε θα δώσω το λόγο για ένα λεπτό στον κύριο Μαριά η έκθεση κονφεράτι δίνει έμφαση σε δύο σημεία πρώτα απ' όλα στην κοινωνική διάσταση της επιχείρησης διότι αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο ιδίως σε μια φάση όπως η σημερινή που αντιμετωπίζουμε μια τεράστια οικονομική κρίση και έχουμε χιλιάδες ανέργους. το δεύτερο είναι η έμφαση στη διαφάνεια διαφάνεια για τη δράση της ίδιας της επιχείρησης διαφάνεια για τις σχέσεις των μετόχων με την επιχείρηση διαφάνεια για το ποιοι είναι οι μέτοχοι διαφάνεια στις σχέσεις των μετόχων με τα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης. πραγματικά σε αυτή τη φάση της παγκοσμιοποίησης υπάρχουν κεντρικά ερωτήματα για ποιο λόγο γίνεται μια επένδυση σε επιχείρηση από πού προέρχονται τα κεφάλαια γίνεται η επένδυση για την ενίσχυση της ίδιας της επιχείρησης ή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή για λόγους φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. επίσης πού πληρώνουν τους φόρους τους οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις; ποιος θα είναι ο ρόλος των ίδιων των εργαζομένων στην επιχείρηση οι οποίοι πρέπει να έχουν ρόλο σημαντικό. σε όλα αυτά απαντάει η έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στην Επίτροπο κυρία Γιούροβα για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Αξιότιμοι βουλευτές, να αντιδράσω εν συντομία στη συζήτηση αυτή για τις εκθέσεις αναχώρα. Να είμαι πολύ σαφής. Συμφωνώ απόλυτα με όλες και όλους εσάς που εκφράσατε την ανάγκη να είναι μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια. Αυτό είναι και προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως βέβαια και πατάξη της φοροδιαφυγής και της φόροαποφυγής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν λέει ναι. Όμως Πρέπει αυτό το πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε με ένα διαφορετικό νομοθέτημα. Είναι η οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων αυτό το εργαλείο. Και εργαζόμαστε με εντατικούς ρυθμούς ε, για αυτό το νέο νομοθέτημα, το οποίο θα εστιάζει ε, εντελώ ε, στη φορολογική διαφάνεια, όπως είπα και προηγουμένως. Επεξεργαζόμαστε κάποια στοιχεία, αναλύουμε ορισμένα στοιχεία για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα κάνουμε προτάσεις που θα αυξάνουν το διοικητικό ε, αλλά αντίθετα θα περιορίζουν τη γραφειοκρατία. Και ελπίζουμε αυτό να το πράξουμε με τον, μεγαλύτερο, με τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο για να έχουμε και τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Χρειάζεται λίγο περισσότερος χρόνος και όπως είπα σχεδιάζουμε να έχουμε μια μελέτη αντικτύπου έτοιμη ε, την άνοιξη του επόμενου έτους. Αυτή λοιπόν είναι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση. Πολλοί από εσάς ε, εκφράσατε την άποψη ότι με την οδηγία αυτή θα αυξηθεί ανταγωνιστικότητα και οικονομική ανάπτυξη. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις απόψεις σας και βασίζομαι ε, στην ε, συνεχή σας υποστήριξη και ελπίζω και να υπερψηφιστεί η έκθεση αύριο. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ την Επίτροπο. Εισηγητήσω και σκοφεράτη για δύο λεπτά τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους που πήραν τον λόγο. Όχι μόνο για όσα είπαν, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο εκφράστηκαν. Η δουλειά που κάναμε ήταν κοπιώδης μακρο, κράτησε πολύ καιρό και έδειξε ότι οι συμβαστικές λύσεις βρίσκονται σε ένα καλό πνεύμα συνεργασίας, πραγματικά αγαστής. Κάτι που δεν ήταν δεδομένο, αλλά το πετύχαμε. Και αυτό πρέπει να αποδοθεί στην καλή διάθεση και την προθυμία και της ε, παιδείας και όλων των σκιωδών και των συναδέλφων που τώρα συμμετείχαν στη συζήτηση. Στόχος μας ήταν αυτός που αναφερόταν και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός που ενισχύσαμε και αναθερμάναμε. Δηλαδή, από τη μια να έχουμε κίνητρα για τους επενδυτές που βλέπουν την εταιρεία ως ένα τόπο που θα παράγει πλούτο και όχι να επιτρέψουμε την κερδοσκοπία. Γι' αυτό η παραμονή ενός ε, μετόχου επενδυτή στην εταιρεία είναι σημαντικό ε, στοιχείο και κίνητρο. Από την άλλη χρειαζόμαστε διαφάνεια, το είπαμε όλοι. Διαφάνεια για να καταπολεμήσουμε την απάτη, τις ανισότητες. Διαφάνεια απλώς και μόνον για να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή και φοροαπάτη το να πληρώνει κανείς τους φόρους είναι καθήκον. Ακόμα και αν για όλους είναι μια θυσία και για τους ε, μεμονωμένους πολίτες αλλά και για μια εταιρεία. Όμως ε, τα κονδύλια αυτά επαναχρησιμοποιούνται για τη σταθεροποίηση και το σταθερό βίο μιας κοινότητας με, μέτρα κοινωνικής πρόνοιας. Γι' αυτό καταβάλουμε το αντίτιμο αυτό. Αυτό είναι αρχή του πολιτισμού και ε, πρέπει να προστατευτεί. Όλοι θα πρέπει να συμμετέχουν στο στόχο για το τελικό αποτέλεσμα. Επίσης για την υποβολή εκθέσεων αναχώρα. Ε, το λέω ε, ιδίω προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Επίτροπο, ότι η έκθεση Καηλή που εγκρίναμε τον Μάρτιο στο Κοινοβούλιο απαιτούσε η υποβολή εκθέσεων αναχώρα να προβλεφθεί μέσω τη άμεση αναθεωρήσεω τη οδηγία για τα λογιστικά στοιχεία. Η οδηγία για τα δικαιώματα επηρεάζει την οδηγία αυτή, οπότε αυτό είναι το σωστό σημείο για να προβλέψουμε αυτό το νέο στοιχείο. Ένα νέο στοιχείο από το οποίο θα εργαστούμε όλοι μαζί, μα σωστό είναι η αφετηρία μα να είναι αυτή. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ τον εισηγητή. Η συζήτηση τώρα